Dear colleague, we can start now. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Sorry. Okay. Allora, we can start now. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σήμερα το πρωί Έχουμε να ψηφίσουμε μία έκθεση και τρεις γνωμοδοτήσεις. Να πάρω κι εγώ την κάρτα μου για να ψηφίσω. Λοιπόν, η πρώτη έκθεση είναι του συναδέλφου Ζαλάτισλαβ Κρασνοντεύσκη που δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα για προσωπικούς σοβαρούς λόγους και Ευχαριστώ τη συνάδελφο Γιάντλιγκα Βιτνέσκα που είναι εδώ μαζί μας και θα διαβάσει μία δήλωσή του εκ μέρους του. Καλώς ορίσατε και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο καθηγητής Κασνοδιεύσκη Κράσνοδιεύσκη ζητά συγγνώμη για την απουσία του απουσιάζει για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πρέπει να βρίσκεται στη Βαρσοβία. Ο καθηγητής ε, Κρασνοντιεύσκη ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες, που ήταν και αρκετοί, και ευχαριστεί και τους ε, σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν ενεργά στην ε, εκπόνηση της έκθεσης ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες ε, σε μεγάλο βαθμό ε, έχουν εγκριθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Καταλήξαμε σε θετικές ε, λύσεις και η έκθεση αυτή Ε, δίνει ε, θετικές ε, υποδείξεις για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσει την Γραμματεία, την Άννα Μαρία Γνωγκέρα και τον Μάρκους Πρέτσια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι έκανε εξαιρετική δουλειά, τη συνάδελφα Σβεντρόβα, ε, Χάνεμπολ, τον κύριο Χουντή, τον κύριο Μαρεγκάλ και ούτω καθεξής και να ευχαριστήσω και εγώ τη γραμματεία. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση, διότι επικαιροποιεί το στρατηγικό πλαίσιο της ε, ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε απάντηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συστάσεων του Συμβουλίου. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να συμβάλλει και το Κοινοβούλιο. Έχω δει ότι υπάρχουν αρκετές συμβαστικές τροπολογίες. Θα κρατήσει αρκετά η ψηφοφορία, επομένως θα ξεκινήσουμε αμέσως. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία 5 του εισηγητή. Ε, υπέρ. nice. <laughs> First morning is <laughs> Είναι νωρίς το πρωί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47. Ε, θέλετε επαλήθευση για την 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Να προσθέσουμε και την ψήφο της κυρίας Χάνιμπολ γιατί είναι σκιώδης συγγήτρια και ξέχασε να βγάλει την κάρτα της. Ακόμα και αν ε, ψηφίσει υπέρ, απορρίπτεται γιατί θα είναι ισοπαλία. Λοιπόν, περιμένω λοιπόν τη μέρη να βρει την κάρτα της, τουλάχιστον για τις επόμενες ψηφοφορίες. Oh Allora, 47. Eh, 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 49. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Όχι, πάμε στη συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Εσείς ψηφίζετε κατά. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Να κάνουμε μια επαλήθευση λοιπόν. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε. 54. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να κάνουμε μία επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ψηφοφορία για την 85 Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Η 84 εγκρίνεται, επομένως περνάμε απευθεία στη συμβαστική τροπολογία 11. Ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά απόχε εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95. Α, επαλήθευση για την 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. 90. Η 94 απορρίπτεται. Εγκρίνεται η 94. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 14 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 του εισηγητέη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται όμως. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, αν θέλετε να το επαληθεύσουμε, αλλά απορρίπτεται, 122 υπέρ, θέλετε επαλήθευση. Είναι σαφές, αλλά τέλος πάντων, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή 1 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά υπέρ συγγνώμη και πάλι κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 19 στην επόμενη σελίδα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, συγγνώμη είναι ταυτόσιμες, δεν ψηφίζουμε, συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Η ισοπαλία. 150 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 152 υπέρ, ...156 πηγαίνουμε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, να κάνουμε μια παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 156. Άρα είστε όλοι κατά, αλλά δεν σκόσετε τα χέρια σας. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 163 του κυρίου Χουντή υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 164 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 189 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 190 που είναι ταυτόσιμο με την 191 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 195 Συγγνώμη, 194 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 190 92 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε μια επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας μπορεί και να εγκρίνεται αλλά εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 95 γιατί εγκρίναμε την 92. Η 95 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 στην επόμενη σελίδα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε 237 ταυτόσημη με την 238, ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 33, υπέρ, είναι απόλυτα σαφής. Τι να επαληθεύσουμε. Συμβαστική τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται, 3, συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, α, συγγνώμη. Είκοσι ένα υπέρ, κα, κατά, αποχές, απορρίπτεται, αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. I go to, uh, Πάμε στην 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Πέραση της ψηφοφορίας. Άρα 22 υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση και πολλά συγχαρητήρια στον εισηγητή και σας, σας βεβαίω που τον αντικαταστήσατε. Ευχαριστώ και όλες και όλους και τους σκιώδεις εισηγητές Ιδίω ευχαριστούμε τον καθηγητή Κρασνοντεύσκη βεβαίω. Τώρα, η δική μου έκθεση. Έχουμε τη γνωμοδότησή μου για την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης για τους πρόσφυγες ε, ε, την ε, ένταξη στην αγορά εργασίας Ευχαριστώ τους και οδησογητές ε, Μάνος ε, Τζαμπάσκι, Μαραγκάλ, Χουντή που συνεργάστηκαν επί του ζητήματος. Βρήκαμε και κάποιες, ε, κάποιους θετικούς συμβιβασμούς και τη συνάδελφο από τη Γραμματεία για την υποστήριξη και τους βοηθούς μου φυσικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας εισακούγεται για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά την ευρύτερη ένταξη χωρίς βέβαια ε, την ε, εκπαιδευτική πολιτιστική ένταξη και την ε, πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, ανώτατης εκπαίδευσης δεν υπάρχει πραγματική ένταξη και το αποδεικνύουν και τα στοιχεία αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία έχουμε συμπεριλάβει είναι πολύ σημαντικά. Ελπίζω να γίνονται και σεβαστές πλήρως οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας από την Επιτροπή Απασχόλησης. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης που προβλεπόταν για τις 5 Μαΐου θα γίνει γίνει στις 30 Μαΐου, άρα εμείς ε, υποβάλλουμε έγκαιρα την γνωμοδότησή μας. Περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία και σας ευχαριστώ και πάλι. One, eh, adopt, ε, Παραγράφος 1, συμβαστική 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14, τροπολογία 14. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, Καλά λοιπόν, ας κάνουμε επαλήθευση. 14. Αρχίζει, λίγη. Εγκρίνεται λοιπόν. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Ψηφοφορία τα τμήματα που ζητούν σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 18. Ζουλό υπέρ, κατά, αποχές. Αυτή απορρίπτεται. 19. Α, με συγχωρείτε, αυτή έχει αποσυρθεί. 21. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα. συμβαστική 4, υπέρ, κατά. Ξανά υπέρ, κατά, ε, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32, κατά τμήματα, ζήτησε το Λαϊκό Κόμμα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36, υπέρ, κατά, απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 53 είναι η πρόταση, υπέρ 43 53 διορθώνει 53 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ αρχίζει 57 πέρας Απερίφθη όπω βλέπετε. 58. Υπέρ. Κατά απόχέ. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά απόχέ Εγκρίνεται. 74. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ υπέρ λοιπόν κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε 76 πάντα τώρα τέλος της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται λέει η πρόεδρος αλλά δεν είναι σωστό ναι, ναι, ναι, ναι, ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 77. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά. Υπέρ πάλι παρακαλώ κατά αποχές 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ας επαληθεύσουμε όμως. Πέρα της ψήφου εγκρίνεται λοιπόν. 101 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3. Η 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4. Υπέρ. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. 3, 4, 5, 6, 1 και 2. Συμφωνείτε. Άρα λοιπόν, ε, όλοι μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία, τέλος, ...24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την συνεργασία σας. Νομίζω ότι δίνουμε μια θετική ε, ένδειξη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περνάμε τώρα στη γνωμοδότηση του συναδέλφου Σδρογεύσκη για την ε, προετοιμασία της μετεκλωδικής αναθεώρησης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου με τη συμβολή του Κοινοβουλίου εν ώψη της πρότασης της Επιτροπής. Να ρωτήσω τον συνάδελφο αν θέλει να πει δυο λόγια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να πω πω δεν υπάρχουν συμβιβαστικέ τροπολογίε, δεν θέλω να το εκλάβετε άσχημα αυτό, η ε, συμβαστικές τροπολογίες δεν χρειάστηκαν έπειτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στην Επιτροπή οι οποίοι εργάστηκαν εξάρτητα από πολιτικές ομάδες για την ε, ε, γνωμοδότηση αυτή. Το Erasmus Plus είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να εμβαθύνουμε στην πολιτισμική πολυμορφία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο Juncker να μας δώσει ε, μεγαλύτερα ωφέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συνενετικότητά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Έχουμε πάντα δύο πολύ σημαντικά θέματα και νομίζω ότι ζητήσαμε πράγματα για τα δύο πιο σημαντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα τρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ίσως, αλλά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ίσως. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος καθυστέρησε. Πέρας. Απορρίπτεται. οκτώ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. εννέα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Με συγχωρείτε. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Όπως ζήτησε το S&D. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εσείς απέχετε. Α, μάλιστα. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Μπορούμε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, νομίζω όμως πως απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 Αντινόλφη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει λοιπόν, περνάμε στην 18. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Δεν εγκρίθηκε. Λοιπόν, 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. «22 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές». Συγχαρητήρια στον Αντρέη Στρογεύσκη και στους κοιόδες εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση ε, του κυρίου Τζαμπάσκη, εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Όπως ε, γνωρίζετε, απουσιάζει. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ο κύριος Τζαμπάσκι είχε μια πτήση στην οποία καθυστέρησε. Σας ευχαριστώ όμως όλους για τη δουλειά και τη στήριξη που του δείξατε. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά, αποχές, παληθεύουμε ηλεκτρονικά, την 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη 14. Πέρας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. 15. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. εκτός μικροφώνου. Επιτρέπετε να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. 50. Χουντής, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. καλύτερα να επαναληφθεί. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ή μπορούμε να προσθέσουμε την ψήφο της συναδέλφου. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, 12 υπέρ, 12 κατά. Λοιπόν, 51. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, Κατά τμήματα ψηφοφορία, όπω ζήτησε το ECR, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 κατά τμήματα, σύμφωνα με το ΕΛΚ, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται πέρας 23 ψήφοι υπέρ καμία κατά 4 αποχές συγχαρητήρια στον συνάδελφο Στρογεύσκη και στους σκιώδεις συζητητές και τη γραμματεία φυσικά. Λοιπόν, τελείωσαν τώρα οι ψηφοφορίες και έχουμε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης παρατηρήσει και συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Σδρογεύσκη για τη στρατηγική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στην προπαγάνδα από τρίτους εις βάρος της. Ο συντάκτης μας λοιπόν θα πρέπει, συγγνώμη ησυχία παρακαλώ, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο κύριε Δρογεύσκη. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα για την Επιτροπή μας. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, να υπενθυμίσω απλώ ότι θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο, μετά θα δώσω πρώτο το λόγο στους και οδησηγητές και από εκεί και πέρα σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για ένα-δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τις και τους συναδέλφους που μου έχουν υποβάλει προτάσεις. Θα αρχίσω με ένα γενικό μέρο, μια γενική παρατήρηση, που είναι σημαντική για την Επιτροπή μας ιδίως. Μα απασχολεί η ρωσική προπαγάνδα και ερχόμαστε να απαντήσουμε σε αυτήν με καθυστέρηση. Η Ρωσία ενισχύει την προπαγάνδα της και προς την Ευρώπη και παγκοσμίως και μάλιστα έχει αρχίσει εδώ και μια οχταετία. Η αντίδρασή μας έρχεται καθυστερημένα. Δεν ε, είναι πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα αυτή με δική μας αντιπροπαγάνδα. Εμείς θα αντιπαρατάξουμε την αλήθεια. Θέλουμε να προσφέρουμε ακριβείς πληροφορίες. Δεν πρόκειται για προπαγάνδα εκ μέρους μας. Θέλουμε να απαντήσουμε στη ρωσική προπαγάνδα παρέχοντας στο κοινό αληθινή γνήσια ενημέρωση. Η κατάσταση ωστόσο δεν είναι απλή δεν πρόκειται μόνο για τα ρωσικά συμφέροντα στην Ευρώπη. Πρόκειται και για αντιμετώπιση άλλων φορέων, όπως για παράδειγμα της προπαγάνδας του ε, Ισλαμικού κράτους. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν την ύπαρξη της ρωσικής προπαγάνδας. Από την άλλη μεριά όμως οι πολίτες μας θεωρούν αναγκαίο να παραμείνουμε προσεκτικοί και συγκρατημένοι. Πού αναφαίνονται οι αποδείξεις ότι λειτουργεί αυτή η ρωσική προπαγάνδα. Ιδίως φάνηκαν στην περίπτωση της προσάρτησης της Κρυμαίας. Επίσης όλες οι πληροφορίες γύρω από την περιοχή του Ντομπάς. Το ίδιο και σχετικά με τραγικά γεγονότα όπως η κατάρριψη του Ολλανδικού τουριστικού αεροσκάφους. Αυτά είναι σημάδια που δείχνουν πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να παραμείνουμε άγρυπνοι και να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για προπαγάνδα από πλευράς τους και όχι απλή ενημέρωση. 60% των Ολλανδών τάχθηκαν στο δημοψήφισμα που έγινε κατά τη σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία. Αυτό το θεωρώ εγώ απόδειξη ότι αποδίδει η ρωσική προπαγάνδα. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έχει ιδρύσει μια ομάδα εργασίας για τα θέματα αυτά. Με σημαντικά θέματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση, σημειώνω και όχι στη γνωμοδοτησή μου απαραίτητα, στην έκθεση μιλούν ιδίω για την ανάγκη στήριξης ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να φροντίσει η Ευρώπη να ενισχύσει τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερο, το έχει επίσης τονίσει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ συμφωνώ. Οφείλουμε να ενισχύσουμε την κατάρτιση των νέων σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει δηλαδή οι νέοι να μπορούν να προσεγγίζουν με κριτικό πνεύμα την ενημέρωση που τους γίνεται. Τρίτο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επιτυχία μας στον χώρο αυτό θα είναι δυνατή μόνο εάν έχει χαρακτήρα μακροπρόθεσμο. Εάν δράσουμε και στο επίπεδο της διπλωματίας και της πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να γίνεται αντικειμενικά και στη βάση της αλήθειας η ενημέρωση από πλευράς μας. Να καταδείξουμε ποιες είναι οι δραστηριότητε μας στην Ευρώπη. Η έκθεση για την οποία μιλούμε σήμερα ε, δείχνει ότι και η δική μας Επιτροπή Πολιτισμού βαδίζει το σωστό δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Τονίζει δηλαδή τα πράγματα που είναι αναγκαίο να τονιστούν. Και στο κάτω τη αυτά δεν έχουν και υπερβολικά μεγάλο κόστος. Ευχαριστώ και για τις αποτελεσματικές προτάσεις σας. Συμφωνώ και για τη διευκρίνηση που κάνατε. Το θέμα δεν είναι να ε, απαντήσουμε στις πληροφορίες αλλά στην προπαγάνδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ε, η κυρία Τζούλι Ward έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ah, sorry. <laughs> Some problem. Uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συντάκτη για τη γνωμοδότησή του. Πρόκειται για ένα πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει πολύ καλά στοιχεία. Για παράδειγμα, την έκκληση για ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ελευθεροτυπία. Ε, το ρόλο της ε, παιδείας ε, και της γνώσης των μέσων ενημέρωσης και να υπάρχει και πολιτιστική διπλωματία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρει λοιπόν πολλά από τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας και καλύπτουμε ως Επιτροπή. Συμφωνώ με τον συντάκτη ότι αυτά θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία θα εδράζεται η γνωμοδότηση από πλευράς της Επιτροπής μας και ως και συγγήτρια θα υποβάλω τροπολογίες προκειμένου να εξελίξουμε περαιτέρω τις ιδέες αυτές και να προσθέσουμε και κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα την ανάγκη να υπάρχει και ένα εναλλακτικό αφήγημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της στρατηγικής της για τα μέσα που θα περιλαμβάνει και ε, συγκεκριμένα στοιχεία βάση περιφερειών και συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων στις χώρες αυτές καθώς επίσης και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τον τοπικό πληθυσμό ιδίω για τους νέους ανθρώπους. Έχω και κάποια πείρα, έχω συμμετοχή σε ε, προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων ε, που δείχνει ε, πόσο θετική μπορεί να είναι η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη της ελευθεριοτυπίας και ανεξάρτητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να υπάρχουν δράσεις υποστήριξης για δημοσιογράφους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται στη φυλακή. Όσον αφορά την ε, γνώση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται διαδικτυακά με τη ρητορία μίσους ε, και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως για παράδειγμα το Twitter και το Facebook. Τέλος, από πλευρά μου θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε περαιτέρω έμφαση στο διαπολιτισμικό διάλογο, επαφές μεταξύ ανθρώπων και ενθάρρυνση της στρατηγικής επικοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συμπεριλάβουμε και τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών. Καμία στρατηγική ήπια δεν μπορεί να επιτύχει ε, εάν δεν υπάρχει πολιτιστική και διπλωματία και διαπολιτισμικός διάλογος και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέραν των συνόρωσης. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις πολιτιστικές ε, ανταλλαγές και κοινωνικές ανταλλαγές ώστε να καταπολεμήσουμε και τις προκαταλήψεις των τοπικών πληθυσμών. Και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και αντιπροσωπείε Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υπεύθυνε για την επικοινωνία στι χώρε εταίρου πρέπει πρέπει να διατηρήσουν και να αυξήσουν κατά την άποψή μου τη μόνιμη επαφή με την κοινωνία των πολιτών και να ε, καταρτίζουν και να επιμορφώνουν καταλήλω το προσωπικό του για να έχουν τι δεξιότητε να τα αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με του κοιόδη ε, συντάκτε και το συντάκτη και θεωρώ ότι το θέμα του πολιτισμού και των ε, μέσων μαζική ενημέρωση τη εξωτερική θέση έχει αποδώσει καρπού και έχουμε έναν οδικό χάρτη για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πολιτιστική Διπλωματία, όπω ανακοίνωσε η Φεντερίκα Μογκερίνη και ο Επίτροπο Ναυράτση την προηγούμενη εβδομάδα στο φόρο Φόρουμ Πολιτισμού εδώ στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην Επιτροπή που εργάστηκαν σκληρά προκειμένου το θέμα αυτό να βρίσκεται ως πρώτη προτεραιότητα και να καταλάβουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι ο πολιτισμός είναι εργαλείο της ήπιας δύναμής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τζούλη. Ο συνάδελφος Uh, well. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας καλωσορίζει μέσα ε, την αγνομοδότηση αυτή και την έμφαση που δίνει ο εισηγητής στην ε, ρωσική προπαγάνδα. Πιστεύω πως είναι πολύ ε, ενδιαφέρον σημείο. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια εάν φταίει η ρωσική προπαγάνδα για την πρόσφατη ψηφοφορία στις κάτω χώρες. Νομίζω πως οι παράγοντες ήταν διαφορετικοί. Όμως η αναφορά στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι εμείς ε, πρέπει να ε, ταχθούμε υπέρ μιας φιλοευρωπαϊκής προπαγάνδας. Πιστεύω πως ε, μια σωστή στρατηγική επικοινωνίας, αντί να τονίζει τα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε ίσως να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης από τη ρωσική πλευρά. Ε, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ήδη κάποια σύγχυση ε, σε κάποιους συναδέλφους σε σχέση με την καταπολέμηση της προπαγάνδας, σε τη διαστολή με την πρόθεση των δικών μας ε, ιδεών για τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πως η γνωμοδότηση θα τύχει μεγαλύτερη στήριξη αν επικεντρωθούμε στον τίτλο, εάν δηλαδή ονομαστεί καταπολέμηση της προπαγάνδας από τη Ρωσία και από τρίτα μέρη. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Μπίλντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση. Παράφως 2. Μιλείτε εκεί για καλά και κακά ΜΜΕ. Ποιος και πότε αποφασίζει ποια είναι καλά και ποια είναι κακά. Δεν έχουμε όλοι την ίδια ερμηνεία. Το κείμενο στρέφεται ιδίω κατά της Ρωσίας όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με την Τουρκία, χώρα όπου δεν ισχύει, δεν πλέον η ελευθεροτυπία. Δεν επέτρεψε για παράδειγμα η Τουρκία την είσοδο σε ανταποκριτή του γερμανικού καναλιού ARD. Επίσης δεν επιτρέπει να λειτουργήσει το Πούτνικ. Αυτά τα έχει καταδικάσει η Γαλλική Ομοσπονδία Δημοσιογράφων γιατί παίζουν το παιχνίδι του Πούτιν. Εγώ ανησυχώ και περισσότερο από την έλλειψη πολυφωνίας και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι διαρκώς, ακόμη και για τους συναδέλφους μου, παίρνουν τα κείμενα και αφαιρούν το όνομά μου. Κάποτε ο Βολτέρος είπε «Δεν συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για να επιτρέπετε να τα λέτε». Και νομίζω ότι αυτή η ρίση έχει και σήμερα άμεση επικαιρότητα. Ευχαριστώ αγαπητή Μπίλτ. Τόμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όλοι μας παρακολουθούμε τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση. καθημερινά. Εγώ έχω μητρική μου γλώσσα τα ρωσικά, γι' αυτό λοιπόν παρατηρώ τον ρωσόφωνο τύπο σε ορισμένε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και είμαι πρώην δημοσιογράφο. Με ανησυχεί η γλώσσα και στα ευρωπαϊκά και στα ρωσόφωνα μέσα ενημέρωση, διότι η πληροφόρηση ειδικά για το θέμα της Ουκρανίας, είχε χαρακτηριστεί από μεροληψία και σύμφωνα με αρκετές στατιστικές, οι Ρώσοι κατά πλειοψηφία δεν εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ένα συστότοπος ρωσόφωνος είναι ε, διαθέσιμος όπου εκεί μπορεί κάποιος να διαβάσει μεταφρασμένα άρθρα από τον ευρωπαϊκό ε, και αμερικανικό ε, τύπο. Αυτός ο ιστότοπος είναι ένα αρκετά χρήσιμο μέσο. Και γιατί, διότι πολλοί ε, Ρώσοι έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν πληροφορίες ανεπηρέαστες από τις ε, ρωσικές επιρροές. Όμως η αποτελεσματικότητα του προγράμματος East Stat δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Και λυπάμαι που το λέω, όμως αυτή εδώ είναι κλασική περίπτωση προπαγάνδας και δυστυχώς ο ρωσόφωνος τύπος είναι φερέφωνο προπαγάνδας. Όμως και εμείς το ίδιο κάνουμε. Πιστεύω πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε μια ουδέτερη και ε, αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, διαφορετικά ε, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης δεν θα καταφέρουν να ανταγωνιστούν τα ρωσικά. Δεν μπορούμε να την καταστήσουμε δηλαδή την προπαγάνδα με άλλη προπαγάνδα. Επίσης πρέπει να καταπολεμήσουμε τη λογοκρισία ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να είμαστε ανοιχτοί στις νέες ιδέες και στις διαφορετικές ερμηνείες ε, μιας είδησης. Τώρα, δυστυχώς η πλήση εγκεφάλου των νέων ανθρώπων ε, υπέρ της τρομοκρατίας δεν φαίνεται στο έγγραφο. Ε, μιλάμε μόνο για τη Ρωσία, αλλά τι γίνεται με το ISIS, τι γίνεται με τον ε, αραβικό τύπο. Πρέπει να ε, δούμε και αυτές τις πτυχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις. Σβεντρόβα στη συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Στρογεύσκη για την γνωμοδότησή του. Όλες και όλοι μας έχουμε τις απόψεις μας. Θυμούμε όμως, διότι διαθέτω τη σχετική εμπειρία, επί 25 χρόνια έζησα σε μια χώρα όπου υφιστάμεθα τότε μαζικά τη ρωσική προπαγάνδα. Και γνωρίζω πόσο επικίνδυνη είναι αυτή. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε τρόπους εργαλεία για να αντιδράσουμε στη ρωσική προπαγάνδα. Θα είναι δύσκολο να επιλέξουμε τα σωστά εργαλεία για να το πράξουμε αυτό και για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποια θα είναι αυτά. Χρειαζόμαστε γνήσια ενημέρωση στη βάση αληθών ισχυρισμών και ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε επίσης για την ε, βράβευση με το βραβείο Lux. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε και το θέμα της πρικοδότησης αυτού του βραβείου. Δεν ξέρω αν αυτό κατάλληλο κανάλι, ωστόσο, για να προωθήσουμε τέτοια θέματα, γιατί το Lux δίνεται για κινηματογραφικά έργα υψηλής ποιότητας. Νομίζω πρέπει να το στηρίξουμε το βραβείο Λουξ για τις ταινίε, γιατί είναι μια από τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες μπορούν να ε, ευαισθητοποιήσουν το κοινό για τις ευρωπαϊκές αξίες. Να μιλήσουμε επίσης με ανεξάρτητες οργανώσεις από την Κρυμαία. Ακούμε ότι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να μιλήσουν με μια ανεξάρτητη φωνή διώκονται ή και εκδιώκονται από την Κρυμαία. Η ρωσική προπαγάνδα είναι ισχυρότατη στην Κρυμαία και οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν καν τον τρόπο να αντιδράσουν και αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν. Εγώ θα στηρίξω λοιπόν την έκθεση. Η κυρία Τρίπελ. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να γίνει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στην προπαγάνδα και την κριτική. Γι' αυτό πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι εύκολο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πιστεύω πως ε, πράγματι υπάρχει ρωσική προπαγάνδα, είναι κάτι που γνωρίζουμε και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις από τον ίδιο τον ε, Πούτιν ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα πρέπει όμως να είναι η απάντησή μας. Θεωρώ πως πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε ότι έχουμε καλές λύσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες, υπάρχει πρόοδος στην επίλυση των προβλημάτων τους. Πιστεύω πως ε, αυτό είναι το πιο πιστικό επιχείρημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να ξεπεραστεί η προπαγάνδα. Τώρα, διαφωνώ με το ότι η ρωσική προπαγάνδα ευθύνεται για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στις κάτω χώρες. Ε, πιστεύω πως υπάρχουν πολλά εσωτερικά ζητήματα τα οποία έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι όντως πολύ σημαντικό η πληροφορία να είναι ανεξάρτητη και ξεκάθαρη, να προωθήσουμε τον ανεξάρτητο τύπο εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλά να κάνουμε και στο εσωτερικό μας, διότι υπάρχει συγκεντρωτισμός και έλλειψη πλουραλισμού σε αρκετές χώρες της Ένωσης. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ενέργειες έτσι ώστε οι πολίτες να ε, απολαμβάνουν ανεξάρτητη, ε, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και πληθώρα πληροφοριών. Γι' αυτό είναι πιστεύω χρήσιμο να στηρίξουμε τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε δημοσιογράφους γειτονικών χωρών να ε, περάσουν ορισμένο καιρό ως μαθητευόμενοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπάρχει και στη ρωσική γλώσσα, αν δεν κάνω Γι' αυτό λοιπόν μπορούν οι ρωσόφωνοι πολίτες να έχουν ε, πρόσβαση σε πληροφορίε σχετικά με το τι κάνουμε. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη η κατάσταση με την ελευθεροτυπία και πιστεύω πως πρέπει να στραφούμε και προ την Τουρκία και τι αραβικές ε, χώρε δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην ε, ρωσική πλευρά. Υπάρχουν πολλές πτυχές τις οποίες πρέπει να, ε, πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις αρκετών των συναδέλφων. Θέλω να σας πω, επειδή έζησα εκείνα τα χρόνια, ο τίτλος της έκθεσης μοιάζει να επαναφέρει ένα ψυχροπολεμικό κλίμα. Η χρήση του όρου προπαγάνδα είναι μια πολύ συζητήσιμη έννοια για να την εισάγει στις σύγχρονες συνθήκες. Όχι πως δεν γίνεται προπαγάνδα από όλες τις πλευρές. Απλώς εδώ ας πούμε στη Δυτική Ευρώπη την λέμε κατεφημισμό επικοινωνία. Προφανώς αυτή η, έκθεση είναι ενταγμένη σε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα που έχει και συγκρουσιακό κλίμα που έχει επέλθει λόγω του Ουκρανικού και όχι μόνο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Προφανώς η Ρωσία έχει τους δικούς της στόχους όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους δικούς της στόχους. Όμως καταλήγω κι εγώ σε ένα συμπέρασμα, σε μια παρατήρηση δεν κινδυνεύει δεν κινδυνεύει, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την όποια προπαγάνδα της Ρωσίας. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε τι να σας πω. Κινδυνεύει από την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πει κάποιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από αλληλεγγύη, από μια πολιτική συνοχής, από μια πολιτική ε, άμβληση των διαφορών μεταξύ των χωρών, από μια πολιτική σεβασμού της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατίας αυτό χρειάζεται να το πει η ρωσική προπαγάνδα. Επομένως, αν κινδυνεύει αγαπητοί συνάδελφοι, η πορεία και η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει από την ίδια την πραγματολογική, την πραγματική κατάσταση. Και επομένως, για κάποιον που θέλει να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, ας δει πώς πρέπει να κινηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ώστε να συγκινεί και να ελκύει τους πολίτες. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, <clears throat> επειδή σχεδόν προσανατολίζεται στο να απαντηθεί η ρωσική προπαγάνδα που υπάρχει επαναλαμβάνω, που υπάρχει επαναλαμβάνω, αλλά ξανασκεφτείτε συνάδελφοι, ιδιαίτερα όσοι είσαστε από, άλλες, ε, από τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, ότι τότε στο ψυχροπολεμικό κλίμα υπήρχε και διαφορετικό στόχο, διαφορετικά καθεστώτα. Τώρα ο Πούτιν λέει ότι είναι και αυτός του δυτικού, του καπιταλιστικού, της ελεύθερης οικονομίας. Άλλο τι κάνει και πώς το εφαρμόζει. Επομένως, ιδεολογικό πολιτικές συγκρούσεις επί της αρχής δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κρατικά συμφέροντα, προφανώς. Άρα, ε, θα έλεγα, η προσπάθεια που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες της να διαδοθούν, να κυριαρχήσουν κτλ. θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις πολιτικές μας και όχι να το ανάγουμε το θέμα σε θέμα προπαγάνδας. Και η τελευταία παρατήρηση είναι και υποκριτική. Εδώ έχουμε προπαγάνδα χωρών από ό,τι συζητούσαμε χτες από την Τουρκία και άλλους κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστολή των ελευθεριών ή περιορισμό των ελευθεριών και, ναι, και εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει αντίδραση. Επομένως ε, αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Φοβάμαι πως είναι μια προσπάθεια για να μετατοπίσουμε το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά είπα τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ να τηρείτε τα δύο λεπτά και όχι παραπάνω γιατί καθυστερούμε. Ο κύριος Βέρ και μετά ο κύριος Δαμάτο. Ευχαριστώ πολύ. Εκπλήσωμαι με όλες αυτές τις ε, συζητήσεις για το θέμα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο για την άποψη αυτή. Πιστεύω πως είναι μία πολύ σωστή άποψη και πρέπει όντως να επιλέξουμε τις σωστές λέξεις για να περιγράψουμε τα σωστά προβλήματα. Το καθεστώς του Πούτιν έχει χάσει ε, το, την ιδιότητα του εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και με τις ε, συγκρούσεις που έχουν... Ε, ε, παρατηρηθεί αυτή τη στιγμή, αλλά έχω να πω ότι η πολιτική της ανατολικής γειτονίας χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια προσέγγισης ε, αυτών χωρών αυτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία προκάλεσε κύματα προσφύγων, νέα κύματα προσφύγων. Πριν από λίγα χρόνια, τα μέσα ενημέρωσης και γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ε, είχαν αυξήσει την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία προσπαθεί μέσω της προπαγάνδας, και πιστεύω πως πολύ σωστά χρησιμοποιήθηκε ο όρος αυτός, να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αποσταθεροποίηση είναι γεγονός. Και αυτό που γράφει ο συνάδελφος εδώ με βρίσκει σύμφωνο. Σε ορισμένα σημεία θα μπορούσε μάλιστα η διατύπωση να είναι και πιο αυστηρή. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις, ε, στο χώρο των δημόσιων επικοινωνιών, αλλά και ε, στην πολιτική. Η επιρροή της Ρωσίας διαφαίνεται όλο ένα και περισσότερο στην ε, πολιτική, με την επιρροή της στις ε, ε, ακροαριστερές ομάδες. Υπάρχουν διαφορές που έχουν παρατηρηθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια. Από τη μία... Η κρίση έχει χωρίσει τα κοινοβούλια σε δύο στρατόπεδα. Άκρο αριστερά, άκρο δεξιά. Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι στηρίζαμε αυτούς που τώρα ε, μας εναντιώνονται. Η ε, κυρία Νταμάτο, να σας συσταθώ. Είμαι νέα στην Επιτροπή και θα συνεχί... ξεκινήσω ως και ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ξεκινάμε λοιπόν τις εργασίες σε αυτή την έκθεση που έχει ως θέμα την προπαγάνδα από τρίτους, κυρίως ε, επικεντρωνόμαστε στη Ρωσία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα πάντα ξεκινούν από ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2015. Επομένως, θα πρέπει λογικά να αποφασίσουμε και βάσει των όσων προβλέπονται από τις συνθήκες. Το άρθρο 21 της συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στον υπόλοιπο κόσμο δημοκρατία, κράτος δικαίου, καθολικότητα και ε, πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, σεβασμό του ανθρώπου και αλληλεγγύη και σεβασμό των Χάρτας των ε, Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει καμία προσπάθεια να απαντήσουμε σε προπαγάνδα ε, έλλειψη νομιμοποίηση από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αντίστοιχη προπαγάνδα που αλλάζει επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στι χώρε μέλη και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε σχέση με τρίτε χώρε. Για παράδειγμα στη διαχείριση περίπλοκων περιπτώσεων όπω για παράδειγμα το προσφυγικό και αναφέρομαι επίση και σε πολύ ευαίσθητε περιπτώσει, ε, όπω για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα των ε, πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Αφρική εις βάρος της αξιοπρέπειας ε, των ανθρώπων. Υπάρχουν πάρα πολύ ευαίσθητα πράγματα, όπως για παράδειγμα αντικειμενικότητα, αντιμεροληψία, ανεξαρτησία αυτών όλων που καλούνται να εκπροσωπήσουν ε, για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και για τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει επίσης να υπάρχει μια συνεπής και πραγματική πραγματική εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξωτερικό επίπεδο ενώπιον των τρίτων τη. Αν δούμε πόσο ε, προβληματικό είναι το θέμα τη κατάσταση τη υγεία, τη ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και τη ενημέρωση σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, πολύ πρόσφατα είδαμε και από το, ε, τους γιατρούς σύνορα πολύ πρόσφατα, το γεγονό ότι ε, προσπαθούμε να δώσουμε μια ειλικρινή ανταπόκριση των γεγονότων είναι πάρα πολύ προβληματικό. Προσπαθώ λοιπόν να συνεισφέρω για να βελτιώσω τη γνωμοδότηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κάποιε διακρίσει ή ανοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε οποιαδήποτε έκφραση ε, κακομεταχείριση, ε, βιαιοτήτων και ε, ε, στέρηση κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων που δεν επιτρέπουν να ζήσει σε κάποιον με αξιοπρεπή τρόπο. Σα ευχαριστώ και καλωσορίσατε ω αναπληρώσατε στην Επιτροπή μα εκ μέρου του EFTD. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η συνάδελφος ε, κυρία Τρούπελ. Πρέπει να προειδοποιήσω και εγώ να μην ε, μετατραπεί η έκθεση σε ένα δικαστήριο που θα δικάζεται η Ρωσία. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετούς. Θεωρώ πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γύρω από αυτήν πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Ε, πιστεύω πως η Τουρκία και ε, το Ισλαμικό κράτος προσπαθούν να ασκήσουν ε, προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωση στην Ευρώπη και εκμεταλλευόμενοι την ελευθεροτυπία αυτό ε, παρατηρείται. Η συνάδελφος κυρία Τρούπελ ε, επέστησε την προσοχή στη σημασία της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και πιστεύω πως έχει απόλυτο δίκιο. Στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει ένας όρος που μπορεί να μεταφραστεί ως ψεύτης τύπος. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης και χρειάζεται πιστεύω να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό. Σίγουρα πρέπει να ενισχύσουμε ε, τις ε, προσπάθειες ε, στήριξη των καλά καταρτισμένων αμερόληπτων δημοσιογράφων. Όμως, όπως υπόθηκε και εγώ διαφωνώ με την ε, αποκλειστική εστίαση της έκθεσης στη Ρωσία. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τις άλλες ε, πτυχές του ε, θέματος. Και εντάξει, το γεγονός ότι υπάρχει ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στα ρωσικά δεν αποτελεί λύση. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει ο ιστότοπος και στα ρώσικα ή στα αραβικά. Αυτό ίσως θα μας έδινε μια δυνατότητα να επιτευχθεί μια κάποια ισορροπία ως προς ε, την πληροφόρηση στις χώρες αυτές, ε, την πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πως πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα και όχι μεμονωμένα. Πολλοί από εμάς ε, ξέρω πως έχουν προσωπικές εμπειρίες με τη ρωσική προπαγάνδα, όμως ας μην περιοριστούμε αποκλειστικά σε αυτό, ας δούμε την γενικότερη εικόνα και σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ Πέτρα. Ε, πολύ σημαντικές οι διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είπε η Πέτρα. Ε, σίγουρα η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη ρωσική προπαγάνδα, αλλά στην ατονιστή ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και να προσπαθούμε να τη διασφαλίσουμε. Ε, το θέμα είναι ότι η προπαγάνδα φορά το μανδύα της ε, ελευθεροτυπίας πολλές φορές. Και με αυτόν τον τρόπο κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα ενημέρωσης, ε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς. Γι' αυτό λοιπόν μας είπε και η κυρία Κάμερ για αυτή την άποψη που επικρατεί στη Γερμανία, ότι ο τύπος λέει ψέματα. και το γεγονός ότι δεν εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις ε, στα μέσα ενημέρωσης συνεισφέρει και σε αυτήν την ε, απώλεια εμπιστοσύνης. Ας δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό μας, ας δούμε τι γίνεται με την ελευθεροτυπία στα κράτη-μέλη, ποιες είναι οι τάσεις, ε, τι συμβαίνει, με τι διαφωνούμε, με τι συμφωνούμε, τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως παραπληροφόρηση ε, και τι ε, ως ε, μεροληψία. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην Ευρώπη να μην δημιουργήσουμε μία δική μας μηχανή προπαγάνδας μια μηχανή προπαγάνδας που θα έχει στηθεί από τις κυβερνήσεις ή κεντρικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θεωρούμε σημαντικό και να το προωθήσουμε. Σημαντικό ε, είναι η ελευθερία του τύπου και αυτό είναι το έργο μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθεροτυπία σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πολυμορφία και την ε, ελευθερία έκφρασης προσωπικών απόψεων χωρίς περιορισμούς. Ας μην περιοριστούμε λοιπόν ε, στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ας δούμε τι γίνεται με τα δικά μας μέσα ενημέρωσης και πώς μπορούμε να τα ε, καταστήσουμε περισσότερο ανεξάρτητα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως, είμαστε, πως χρειάζεται να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι δεν πρέπει να επιτρέπεται σε μια δημοκρατική Ευρώπη. Χρειάζεται πληροφόρηση, αντικειμενικότητα, πολυμορφία για τους πολίτες, διότι μόνο έτσι οι πολίτες θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων τους. Ευχαριστώ για αυτή την επισήμανση. Ε, θα πάρω και εγώ το λόγο αργότερα, ο συνάδελφος Βέντε, και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σδρογεύσκη που αναφέρθηκε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό και ε, το γεγονός ότι προσπαθεί να βρει και μια λύση η παρουσίαση των πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, δείχνει λίγο την κατάσταση και ε, καταδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε και λίγο επικριτικοί με τον τρόπο που παρουσιάζονται. Πρέπει να δούμε και το θέμα του προπολογισμού. Η κυρία Τρούπελ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για τους πολίτες ως ένα στοιχείο κλειδί προκειμένου να παρουσιάσουμε την ιστορία μας στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη, κυρίως για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε αυτές τις ανεξάρτητες πληροφορίες. Πολλοί χρησιμοποιούν τον όριο ο μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάποιοι αναφέρονται σε εθνικά μέσα ενημέρωσης. με τον τρόπο αυτό χάνονται πάρα πολλές από τις κοινωνικέ ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζονται κάποια πράγματα. Έχουμε και μία παρουσίαση, για παράδειγμα, της πραγματικότητας του προσφογικού ζητήματος και ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης, οι πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν με ένα αρνητικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν αυτά τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να δίνονται κατάλληλες και οι πιο εύστοχες πληροφορίες, ώστε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βλέπουν λίγο με πιο κριτικό βλέμμα τα όσα παρουσιάζονται. Και εγώ νομίζω ότι ε, και στα αθλητικά κανάλια ε, με κάποιο τρόπο γίνεται προπαγάνδα με τον τρόπο που παρουσιάζονται πληροφορίες. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις πιέσεις έξωθεν. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της για τη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν θα θέλαμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εδώ για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που εκπροσωπείται εδώ από τον συνάδελφο Καλένσκι από την ε, ε, Task Force, την ομάδα Ινδικών Καθηκόντων Ιστάτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμενε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας τη Ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, η αξιολόγηση που έγινε από τους ομολόγου μας είδαμε ότι πρέπει, έδειξε ότι πρέπει να υπάρχουν ε, δυνατότητες για καλύτερη κατανόηση της κοινή γνώμης ε, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εκστρατείες οι οποίες θα προωθούν τα ωφέλη της μεταρρύθμισης. Υπάρχει στήριξη από διάφορα μέσα χρηματοδότησης, όπως το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Μέσο Σταθερότητας. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι τα θέματα τα οποία σχετίζονται με μέσα ενημέρωσης μπορούν να αποτελούν το βασικό στόχο, στόχο ή κάποια από τις συνιστώσεις των προγραμμάτων. Επίσης, πρέπει να προωθήσουμε την πολυφωνία των μέσων και την ελευθερία των μέσων, να υποστηρίξουμε δεξιότητες και επαγγελματισμό τους δημοσιογράφους, ε, να υποστηρίξουμε δημόσια δίκτυα ε, και επίσης να προωθήσουμε ε, δεοντολογικά πρότυπα μέσων ενημέρωσης και διάφορες πρωτοβουλίες των μέσων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι ήδη εν εξελίξη και μέσω των αντιπροσωπιών τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξη προς δημοσιογράφους ε, για δημοσκοπήσεις και παρακολούθηση των μέσων και ε, κατάλληλη νομοθεσία των μέσων. Στην Ρωσική Ομοσπονδία υπάρχουν προγράμματα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να παρουσιάζεται τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Αυτό καλύπτει τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Επίσης, χρηματοδοτούμε ε, δράσεις δημόσιας διπλωματίας που παρουσιάζουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες σε think tank ε, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό στη Ρωσία. Τώρα, για το ανοιχτό πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία του τη πολυδοσκόπηση και του προβληματισμού. Θα ξεκινήσει με 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δύο βασικά θέματα ε, επικοινωνία, ε, ανατηλική και νότια γειτονία και καλύπτει εκστρατείε ενημέρωσης και επικοινωνία. Η Ρωσία δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογή, αλλά οι πληροφορίες που δίνονται θα είναι διαθέσιμες και στη ρωσική γλώσσα. Επιπλέον, το Open Program χρηματοδοτεί το λεγόμενο Media Hub που υποστηρίζει δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, για τα όσα γράφουν και παρουσιάζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε οπτικοακουστικά προγράμματα και θα υπάρξει εκπαίδευση πάνω, άνω των 700 δημοσιογράφων και θα υπάρχουν και ε, σημαντικά προγράμματα και ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης θα μπορούσαν να συμμετέχουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι και ε, εργαζόμενοι στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δημιουργίας ικανοτήτων και θα υποστηρίξουμε και τους ε, managers ε, των μέσων ενημέρωσης αυτών και θα καλύπτουμε και ένα δίκτυο δημοσιογράφων ως μέσο βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφορών και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί και μετά το πέρας του προγράμματος. Θα είναι μια πλατφόρμα για την ε, παρουσίαση περιεχομένων σε διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ρωσικά. Επίση, θέλουμε να διευκολύνουμε ανταλλαγέ ε, μεταξύ επαγγελματιών και βέλτιστες πρακτικέ, ε, υποτροφίε για φοιτητέ και νέου επαγγελματίε που χρηματοδοτούνται από το Erasmus Plus και το Ευρώπη 2020. Θα υπάρχει επίση ε, διαδικτυακά μέσα ενημέρωση, μεταδόσεις μέσω ενημέρωση, εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούμε για να διαβιβάσουμε τα μηνύματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δραστηριοτήτων τη στην γειτονία. Grazie per questo importante Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις σημαντικές διευκρινήσεις. Πριν δώσω το λόγο στο συντάκτη, θα ήθελα να επισημάνω και εγώ κάποιες πτυχές που θεωρώ σημαντικές, ώστε η γνωμοδότηση αυτή να ε, περιλαμβάνει όλα τα πιθανά προβλήματα και την κατάλληλη ισορροπία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Ε, και ακούσαμε πολλά πράγματα από του συναδέλφου. Καταρχά, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διευκρινήσει που είναι πολύ σημαντικέ. Εμεί γνωμοδοτούμε επί τη έκθεση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επομένω, είμαστε στη πλαίσια τη πολιτική γειτονία και τη ε, στρατηγική επικοινωνία τη. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε εμπειρίε στο παρελθόν, αλλά πάντα είπαμε ότι αυτά όλα πρέπει να τα ενισχύσουμε προσπαθώντας να ενισχύσουμε και την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μεταξύ δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης στις χώρες γειτονίας. Σημαίνει ανατολική γειτονία, αλλά και νότια γειτονία και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από το συντάκτη να λάβει υπόψη του και ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, διότι ε, και εσείς είπατε προηγουμένως ότι ένα από τα αιτήματα που είχατε ήταν να υπάρχουν ε, δυνατότητες αυτή η νέα πλατφόρμα να παρέχεται και στα ρωσικά και στα αραβικά ε, και αυτό είναι απάντηση στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τη γειτονία με ολιστικό τρόπο. Υπάρχουν πολύ σημαντικές εμπειρίες ε, και στα πλαίσια της δημιουργίας θεσμικών οργάνων, εκδημοκρατισμού, παραδείγματος χάρη, το EBU το ε, κανάλι μετάδοσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξέπεμπε στην Τινησία ε, και στον Αραβικό κόσμο μετά τις πρώτες εκλογές. Τώρα πιο πρόσφατα υπήρχε και μια συνεργασία με τα δημόσια κανάλια και οι δημοσιογράφοι αυτών των καναλιών ορισμένες φορές χρησιμοποιήθηκαν για προπαγάνδα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας των μέσων ενημέρωσης και μεγαλύτερες σχέσεις με την Ευρώπη. Βλέπω ότι χρησιμοποιείται και το Erasmus Plus και το ορίζοντα, τον ορίζοντα 2020, αλλά νομίζω ότι στη νέα διπλωματία πολιτισμού που προσπαθεί να προωθήσει, είπατε εκπρόσωπος Μογκερίνη, μαζί με τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα πολιτισμού και τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα συνεργασίας, είναι πολύ σημαντικά γιατί πρέπει να βρούμε επιπλέον πόρους και θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής συνεργασίας και ασφάλειας πέραν των εξωτερικών σχέσεων. Αυτές οι επενδύσεις είναι σημαντικές και γι' αυτό. Δεύτερον, Πολύ σωστά είπαν αρκετοί συνάδελφοι ότι πρέπει να έχουμε κατά νου όσον αφορά την Επιτροπή μας, όπως ε, είπε και ο συνάδελφος Ντροβιέσκη σε μία από τις παρατηρήσεις του, να εξετάσουμε και τα εσωτερικά μας ζητήματα. Η προπόθεση για να είμαστε εμεί αξιόπιστοι, όπω είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, συνάδελφο Αμάτο, συνάδελφο Τρούπελ και άλλοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι συνθήκες πολυφωνίας ε, ελευθερίας έκφρασης και έλλειψη συγκεντρωτισμού και εκφοβισμού των δημοσιογράφων ε, θα πρέπει να γίνεται και στα εσωτερικά μας θέματα. Έγινε και μια συνάντηση και εκ μέρους της Επιτροπής μας αλλά και εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας καλέσαμε το παρατηρητήριο πολυφωνίας ε, των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη που εδρεύει στη Φλωρεντία και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και ευαίσθητες οι καταστάσεις ε, και πρέπει λοιπόν να τις υπενθυμίσουμε. Και κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και το γεγονός ότι η προπαγάνδα εντό εισοδηγικών ή τέλος πάντων μία παρουσίαση η οποία δεν ομοιάζει καθόλου και έχει πολλά αλλαγμένα στοιχεία της πραγματικότητας της Ευρώπης αυτή τη στιγμή ε, είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται και οι ξένοι μαχητέ για ριζοσπαστικοποίηση και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε μόνο προς μία κατεύθυνση, πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα, πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα και να μαθαίνουμε και από τους συναδέλφους. Θα λέω ότι συνάδελφοι γιατί και εγώ δημοσιογράφος ήμουν αρχικός. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν της συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να ε, επικοινωνεί η ίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με από τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα και είναι πολύ σημαντικό να το επενθυμίσουμε αυτό. Να ευχαριστήσω τους αδέλφους που έλαβαν το λόγο. Είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ο συντάκτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας κρύψω ότι αντιμετωπίζουμε όντως ένα πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα δεν θα υπήρχε και η γνωμοδότησή μου. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ε, επιθυμώ να τονίσω ότι η προκείμενη γνωμοδότηση γίνεται λόγω εκθέσεως που συντάσσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έτσι δεν είναι. Η δική μας νομοδότηση προβάλλει βεβαίως μόνο απόψεις μας οι οποίες ε, άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Δεν μπορούμε να πούμε σε αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Πρώτο, ο τίτλος και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν. Στον τίτλο μιλούμε για τρίτα μέρη, για τρίτους, δεν μιλούμε για τη Ρωσία ειδικά. Στον τίτλο Μιλούμε για μέτρα που λαμβάνουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρίτη. Άρα εδώ υπονοούνται και η Τουρκία και ενδεχομένως αραβικές χώρες ή άλλες χώρες. Τρίτο, πρέπει να εξετάσουμε την έννοια προπαγάνδα. Η προπαγάνδα δεν σημαίνει μοναχά λάθος πληροφορίες, ψευδείς πληροφορίες, γιατί κάτι τέτοιο θα την έκανε αποτυχημένη. Η προπαγάνδα μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο εάν αναμειγνύει αληθείς, γνήσιες πληροφορίες με μη αληθείς. Δεν αναφερόμαστε στη γνωμοδότησή μου, δεν θα πρέπει να αναφερθούμε μονάχα σε αναλήθειες που προβάλλει η ρωσική προπαγάνδα. Ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται από τρίτους δεν χρειάζονται αντίμετρα δικά μας. Αυτό είναι σωστό. Θέλω ωστόσο να έρθω σε δύο συμπληρωματικά θέματα. Θα συμφωνήσω με μία συνάδελφό μου που τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Χρειαζόμαστε τέτοιες ιστοσελίδες που μπορούν να ενημερώνουν ανθρώπους στη γλώσσα τους και πρέπει να αντιταχθούμε... και στα κηρύγματα μίσους, ιδίως αυτά που προβάλλονται μέσω του διαδικτύου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τις δικές μου παρατηρήσεις προκύπτει ότι αυτή η ρητορική του μίσους λαμβάνει πλέον επαγγελματικό χαρακτήρα. Βγαίνει από μια εσωτερική επιθετικότητα, πολλές μορφές όμως των κηρυγμάτων αυτών μίσους αρχίζουν να παίρνουν ένα χαρακτήρα επαγγελματικό. Αυτά τα επαγγελματικά εντό αγωγικών κηρύγματα μίσους πρέπει να μας απασχολήσουν. Αποτελούν πολύ μεγάλη πρόκληση σήμερα. Αυτά τα κηρύγματα μίσους, επαναλαμβάνω, παίρνουν πλέον χαρακτήρα επαγγελματικό. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα. Δεύτερο ε, θέμα, πολύ σημαντικό. Στην υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας της Επιτροπής Εξωτερικών μιλούν συχνά για υβριδικό πόλεμο. Έχουν ορίσει τι σημαίνει ο υβριδικό πόλεμο. Δεν επιτρέπεται να λησμονούμε όμως ότι σε αυτού του είδου τον πόλεμο πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η προπαγάνδα. Υπάρχουν τελικά στρατιωτικά τμήματα στον Ντομπά ή όχι. Υπάρχουν αυτά τα εντό εισαγωγικών πράσινα ανθρωπάκια, ναι ή όχι. Πώ θα χαρακτηρίσουμε την προσάρτηση τη Κρυμαία, πρόκειται για γνήσια προσάρτηση, πρόκειται για κάτι άλλο. Εγώ έχω δηλαδή αναφερθεί εδώ και στην γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και εγώ έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και επαγγελματικά στο παρελθόν. Έχω να επισημάνω ότι η ρωσική προπαγάνδα δεν θα ήταν επιτυχής εάν δεν είχε τα στοιχεία που σας έχω ε, εξηγήσει ήδη. Τώρα έρχομαι στο Ολλανδικό δημοψήφισμα. Δεν υπήρξε μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν υπήρξε μόνο αποτέλεσμα προπαγάνδας. Βεβαίως η προπαγάνδα έπαιξε ένα ρόλο. Η έκβαση του δημοψηφίσματος είναι βεβαίως περίπλοκη. Δεν υπάρχει θέμα, το αποτέλεσμα έχει ένα περίπλοκο χαρακτήρα. Και ακόμη δύο ε, θέματα. Δεν επιτρέπεται να λησμονήσουμε ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη γλώσσα. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε κριτικοί αλλά να δείχνουμε και ανεκτικότητα και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και μια ανθεκτικότητα απέναντι στην προπαγάνδα, ιδίως μεταξύ των νέων. Πρέπει να αναπτυχθεί το κριτικό πνεύμα των νέων, ιδίως. Ωστόσο, πάντα μέσα στα όρια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, αφού έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα, το οποίο βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Στροβιέφσκη. Κυρίω αυτό το θέμα τη παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση, την οποία θα ε, παρακολουθήσουμε από πλευρά σκιωδών, ε, εισηγητών. Η Επιτροπή Πολιτισμού ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 2 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο. Να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Στέφανο Μαούλου έχει αναλάβει το θέμα αυτό, τον ε, συγχαίρω και το εύχομαι καλή τύχη γιατί είναι το πρώτο θέμα που αναλαμβάνει για την ε, ε, συχνότητα 470-790 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κοινό πλαίσιο προκειμένου να είναι αποτελεσματική η χρήση ε, των συχνοτήτων και να υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές για τα ευρυζωνικά δίκτυα και να προβλέπει και κάποια μέτρα συντονισμού στο μεταβατικό στάδιο. Η έκθεση αυτή ασχολείται με το θέμα αυτό, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι Η πρώτη πρόταση έλεγε ότι πρέπει να γίνει η κατανομή μέχρι τον ε, Ιούνιο του 2016. Ε, ε, ο εισηγητής φυσικά θα υποστηρίζετε και από τους κοιόδης εισηγητές, ε, κυρία Κάμερβεντ, ε, Τρούπελ κλπ. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία που θα εργαστεί επί του ζητήματο. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει ιδιαίτερα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από πλευράς Επιτροπής γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, τι θα γίνει με αυτό το τμήμα τη ε, ζώνη συχνοτήτων γιατί είναι πολύ σημαντική για τι επικοινωνίε, ε, αλλά και για την τηλεόραση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μαούλου για να παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μια σύντομη εισαγωγή επισημάνατε πόσο σημαντική είναι αυτή η γνωμοδότηση σε σχέση με τα όσα ήδη μα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τη τηλεόραση περιλαμβάνει και τι συχνότητε που αναφέρεται από το 470 μέχρι τα 790 MHz. Να υπενθυμίσω σε όλου ότι υπάρχει συνεχή ζήτηση για ευρυζωνικέ ασύρματες υπηρεσίες και mobile data, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολλέ πιέσει για τη δυνατότητα των δικτύων αυτών και επομένω υπάρχει συνεχώ ζήτηση για περισσότερε συχνότητε. Η Επιτροπή μας θα ασχοληθεί με τα θέματα. Θέλουμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και ε, στα 700 MHz η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα ε, κοινό πλαίσιο για να είναι διαθέσιμη αυτή η συχνότητα για τα ευρυζωνικά δίκτυα με βάση εναρμονισμένες τεκτικές ε, και υποστήριξη κατάλληλη για τη μετάβαση. Τα 700 MHz ε, θα πρέπει να δοθούν στα ασύρματα δίκτυα το αργότερα μέχρι το 30 Ιουνίου του 2020. Παρακαλώ λίγο πιο αργά αν μπορείτε. Κάτω από τα 700 MHz ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει μια μεγαλύτερη προθεσμία, πιο μακροπρόθεσμη για οπτικοακουστικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση του ραδιοφάσματος για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τα διαφορετικά επίπεδα της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων θα είναι διαθέσιμη κατά προτεραιότητα για τις τηλεοπτικές υπηρεσίες αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και μια επιλογή ευελιξίας και προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι συχνότητε αυτές και σε άλλες υπηρεσίε, υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Ο συντάκτης της νομοδότησης εκτιμά με τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη του και τι συγκεκριμένε ανάγκες για τα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει για τρία θέματα ουσιαστικά. Η προθεσμία για τα ζώνη των 700 MHz και τη μετάβαση σε ε, ε, ευρυζωνικά δίκτυα είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση, ιδίω ε, για όλες τις χώρες τις οποίες η επίγεια ψηφιακή, ψηφιακή τηλεόραση είναι η βασική πλατφόρμα για την μετάδοση των τηλεοπτικών καναλιών. δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ομογένεια. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη ε, προκηρύξει διαγωνισμό για τα 700 MHz, ενώ η Σουηδία και η Φιλανδία έχουν ε, προγράμματα για την ανακατανομή των ραδιοσυχνοτήτων τα επόμενα χρόνια. Τα περισσότερα όμω κράτη-μέλη έχουν δώσει άδειε ε, στα 700 MHz για μετάδοση, οι οποίε είναι πέραν του 2020. Επομένως, Μία πολύ αυστηρή προθεσμία για την απολευθέρωση της συχνότητας των 700 MHz από, τα τηλεοπτικά, ε, από τις τηλεοπτικές συχνότητες, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020, σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να έχουν αυτό το μεταβατικό διάστημα το οποίο θα χρειάζονται σίγουρα. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την αυστηρότητα, ο εισηγητής προτείνει να πάμε στις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Επίση, προκειμένου να μπορέσουμε να εγγυηθούμε σε όλα τα κράτη-μέλη ότι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσουν να διαθέσουν τη συχνότητα των αυτοχωσίων MHz ε, για τι κινητέ υπηρεσίε, ε, θα πρέπει ε, να λάβουν υπόψη και τα όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση ΛΑΜΗ. Δηλαδή, αυτό το οποίο χρησιμοποιεί και ως μπούσιλα ο εισηγητής. η δυνατότητα να υπάρχουν τεχνολογίες κάτω των 700 MHz, ε, το να υπάρχουν ε, λοιπόν ε, και δυνατότητα σύρμα των ευρυζωνικών δεχνίων αλλά και τηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως πρότεινε και η ομάδα εργασίας για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην γνωμοδότησή της το 2015, πρέπει να καθορίσουμε ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου κάτω των 700 MHz και από τα 570 ε, μέχρι τα 640 MHz και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε μέχρι τα 2030. Ο εισηγητής λοιπόν θεωρεί ότι εδώ δεν χρειάζεται ευελιξία, προτείνει να ε, διαγραφεί αυτό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4 της πρότασης. Κάτω των 700 MHz θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συχνότητα για τα τηλεοπτικά προγράμματα μέχρι το τέλος του 2030, όπως προβλέπεται και στο πρώτο άρθρο παράγραφος 6α και να γίνει μια εξέταση το 2025. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή την εναλλακτική λύση και να προβλέπουμε μόνο μακροπρόθεσμη αλλαγή, εάν είναι συμβατή με τις μεταδόσεις που κάνει το κράτος μέλος και τι κατανομή κάνει το κράτος μέλος στο ραδιοφάσμα και λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες που υπάρχουν πρέπει να έχουμε εκθέσεις προόδου το 20, το 25 και το 30 και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πολύ σημαντικό θέμα του κόστους ε, της ε, μετάπτωσης και των παρεμβολών. Ε, συχνότητα των 700 MHz ε, και η αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και τεχνικές μετατροπές επειδή αλλάζουν οι συχνότητες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αλλάξουν και τις συσκευές που χρησιμοποιούν και θα πρέπει να γίνουν και τροποποίησεις στις υποδομές. Όλα αυτά σημαίνει ότι θα υπάρχει ε, σημαντική επιπλέον επιβάρυνση. Από την εμπειρία που κάναμε με την αλλαγή των 800 MHz, ε, διαπιστώσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν παρεμβολέ ε, στι ε, γειτονικέ συχνότητε. Επομένω, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση θα προστατεύεται, ε, κυρίω και για την αξία που έχει από πλευρά μετάδοση πολιτισμικού περιεχομένου και την άμεση, έμεση σχέση που υπάρχει με τι σχέσει εργασία. Ε, γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε ε, τα κράτη-μέλη εγκαίρως να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους για να γίνει η μετάπτωση και επίσης ε, να δούμε και τι γίνεται για να μειώσουμε τις παρεμβολές ε, με τις υπηρεσίες μετάδοσης. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να αποφύγουμε παρεμβολές από τη χρήση των ασύρματων δικτύων στα τηλεοπτικά δίκτυα και τι γίνεται κάτω από τα 694 MHz. Γι' αυτό είχαμε το άρθρο 5. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι προσπαθούμε να εξετάσουμε τα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν με την ανακατανομή ε, και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, αλλά φυσικά σε καμία περίπτωση εις βάρος ε, του ρόλου που διαδραματίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια και ε, της ε, δημόσιας κυρίως τηλεόρασης. Να δώσω τώρα το λόγο η κυρία Καμερέβερ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, καθώς επίσης ευχαριστώ τον συνάδελφο Μαύρο Πράγματι, εξαιρετική έκθεση. Τον εννοώ τον κύριο Μαλούλου βέβαια. Την υποστηρίζω απόλυτα. Ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Ο συνάδελφός μου έχει περιλάβει όλα τα σημαντικά θέματα της Επιτροπής Πολιτισμού. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που παραπέμπει και στην έκθεση Λαμή που είναι μια πραγματικά ισορροπημένη πρόταση για την πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνώ με την διαγραφή της ρήτρα ευκαμψίας από την πρόταση που θεωρώ ότι όπως ήταν διατυπωμένη ανοίγει πόρτες και παράθυρα στις χώρες μέλη ώστε αυτές να μπορούν να αφαιρέσουν συχνότητες από τους ραδιοσταθμούς εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητες για αυτούς. Πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και για τα θέματα και για, το κόστος μετακίνησης. Έχουμε και τις ε, σχέσεις, έχουμε και τις, ναι. τις των συχνοτήτων δηλαδή. Έχουμε τις σχετικές εμπειρίες λοιπόν ότι δηλαδή το κόστος της μετάπτωσης αυτής δεν είχε αναλυφθεί ούτε καλύφθηκαν από τα έσοδα από τις δημοπρασίες. Ίσως κάποιος μεγάλος ραδιοσταθμός έστω και με δυσκολία να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει αλλά υπάρχουν πολλές μικρές θεατρικές οργανώσεις οι οποίες αναγκάστηκαν να χάσουν τις συχνότητές τους αυτές χωρίς να έχουν καμιά αποζημίωση διότι οι χώρες μέλη δεν είχαν θεσπίσει τις σχετικές ρυθμίσεις. Να προβλέψουμε λοιπόν υποχρέωση των χωρών μελών για την αποζημίωση για το κόστος αυτό. Εμείς το είχαμε συζητήσει ως Επιτροπή Πολιτισμού και εν προκειμένου πρέπει και σαφώς αλλά και, με, και ενωμένοι να ασκήσουμε πίεση στην Επιτροπή Ήτρε. Θυμούμε μακρές και εντατικές συζητήσεις στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία όταν η Επιτροπή Βιομηχανίας μας είχε, είχε προσπαθήσει να μας πείσει τότε, δεν και καλά, ότι τηλεόραση θα βλέπει πια ο κόσμος μόνο μέσω διαδικτύου και όχι με τον ε, τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα, με αναμετάδοση, χερσαία αναμετάδοση δηλαδή. Γι' αυτό θα χαρώ, εάν μπορούμε, όπως είπα, ενωμένοι με μια φωνή ως Επιτροπή Πολιτισμού απέναντι στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Δεν ξέρω αν η στάση τους θα είναι τόσο έντονη όπως την προηγούμενη θητεία, ελπίζω όχι, αλλά πάντως πρέπει να βρούμε κάποια λογική μορφή συνεργασίας με την Επιτροπή Βιομηχανίας. για να επιτραπεί να συνεχίσει η λειτουργία των χερσαίων ραδιοσταθμών. Το μόνο σύστημα μετάδοσης που χρειάζεται να εξασφαλίσει το μέλλον του, ώστε μέχρι το 2030 να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να εκπέμπει στο εύρο συχνοτήτων κάτω από τους 700 ε, μεγάκυκλους. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να μας απασχολήσει και να διαθέσουμε και τα σχετικά κονδύλια. Πολύ σημαντικό αυτό για να διατηρηθεί η πολυφωνία απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό βέβαια το διασυνδέω με το ζήτημα που μόλις συζητήσαμε προηγουμένως. Θα χρειαστεί να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για την έκθεση, αλλά πολύ λίγες, διότι όπως είναι, είναι σχεδόν απόλυτα εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς κυρία Τρίπελ. Με συγχωρείτε, όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ε, όχι εσείς, όχι εσείς. Η κυρία Τρίπελ τελικά. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ με τη γραμμή του, με τη γραμμή που προτείνει. Νομίζω ότι έχει περιλάβει όλα τα βασικά και η κυρία Κάμερ Εβερτ είπε πράγματα που βρίσκω σωστά. Θέλω να τονίσω ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ξανά και ξανά ότι ενισχύεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε εκείνους που χρησιμοποίησαν έως τώρα τις συχνότητες και προσπαθούν να τις διατηρήσουν στην στη χερσαία ε, ραδιοφωνία και στην κινητή τηλεφωνία και, άλλες σχετικές, ε, και άλλους σχετικούς κλάδους προσπαθούν να αποκτήσουν όλο και περισσότερε συχνότητε. Οι συχνότητε είναι δημόσιο αγαθό και αυτό είναι κέριο σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί ξανά στην ε, παρούσα έκθεση. Είπε, Πέτρα, πριν ότι αυτό το σύστημα το, της χερσαίας μετάδοσης είναι κοινόχρηστο, είναι κοινό αγαθό. Και επομένως και η τεχνική υποδομή παίζει και ένα ρόλο. Θα χρειάζεται λοιπόν κάποια προσοχή εδώ. Τώρα γνωρίζουμε επίσης ότι σε ορισμένες χώρες έγιναν οι δημοπρασίε για τις ε, συχνότητε μέχρι τους 700 ε, μεγάκυκλου. Όχι όμως σε όλες. Χρειάζονται λοιπόν και κάποιες μεταβατικές περίοδοι, διότι η χερσαία αναμεταδόμενη τηλεόραση εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλέ χώρε μέλη. Και αυτό θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν πρέπει λοιπόν να τεθεί σε κίνδυνο. Γι' αυτό συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Μαλούλου. Η ε, ρήτρα ευκαμψία δηλαδή που ήθελε να εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σωστή και δεν έχει έρθει ο χρόνο για να γίνει. Σωστά μίλησε και για την έκθεση Λαμή. Μετά το 2030 θα πρέπει να ανοίξει το εύρο συχνοτήτων και από το Δεκέμβρη του 2022 να ανοίξει για νέες υπηρεσίες το εύρο συχνοτήτων μέχρι τους 700 ε, MHz. Δεν χρειάζεται λοιπόν περιττή πίεση ούτε περιττή ανασφάλεια για ε, την ε, χερσαία αναμεταδεδόμενη τηλεόραση και ραδιοφωνία. Άλλο θέμα στις προτάσεις του κ. Μαλούλου είναι το ερώτημα δηλαδή εάν εξετάσουμε ξανά την χρήση των συχνοτήτων. Είχε προτείνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 749 μεγακύκλους, να σταματά εκεί δηλαδή. Η πρόταση γίνεται τώρα όμως να φτάσει μέχρι τους 960 για τις, τις νέες υπηρεσίες δηλαδή. Άρα να ανοίξει ένα ολόκληρο εύρος χρήση των συχνοτήτων. Αυτό μου φαίνεται σωστό ως προσέγγιση. Και από τη δική μου πλευρά λοιπόν ελάχιστες τροπολογίες θα υποβάλω Νομίζω ότι για την Επιτροπή Πολιτισμού το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πώς θέλουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο τρόπο την πολιτική συχνοτήτων τα επόμενα χρόνια και πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται βεβαίως στην Επιτροπή Ήτρε. Χρειαζόμαστε επιχειρήματα για να συμπαραταχθούν μαζί μας ε, τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να διασφαλιστεί ότι η χερσαία αναμεταδεδόμενη ραδιοφωνία έχει μέλλον, τουλάχιστον μέχρι το 2030. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά σε ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα. Πολλές φορές αυτά τα τεχνικά ζητήματα είναι και τα σημαντικότερα. Γι' αυτό λοιπόν συγχαρητήρια για το θάρρος που δείξατε στην ανάληψη ενός τόσο δύσκολου θέματος. Πολλές φορές ως συντονιστής της ομάδας SCR e αναλαμβάνω τέτοιου είδους εκθέσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το θέμα. Ένα από του λόγου είναι ότι η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση είναι, όπω γνωρίζουμε σε αυτήν την επιτροπή, η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα επικοινωνία. Φτάνει σε πάνω από 400 εκατομμύρια νοικοκυριά και για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι όλοι οι σταθμοί, το BBC1, 2, το ITV, το κανάλι 4 και το κανάλι 5, δημόσια τηλεόραση δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτέ τι συχνότητε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, διασφαλίσουμε η ομαλή μετάπτωση στο, στις συχνότητε συχνότητες χωρίς να επηρεάσει την πρόσβαση των καταναλωτών στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Ε, η τεχνική μετάπτωση λοιπόν θα απαιτήσει πολλέ αλλαγέ και αποτελεί πρόκληση ίδια για πολλά κράτη-μέλη. Η ομάδα ECR λοιπόν στηρίζει με την ε, ε, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απελευθερώσει το ευρώ συχνοτήτων το συντομότερο δυνατόν, όμως πρέπει να επιτρέψει κάποια ευελιξία ε, και να είναι ανεκτική στις καθυστερήσεις. Ενδεχομένως θεωρούμε πως θα χρειαστεί περισσότερος καιρός έτσι ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η μετάπτωση. Η ομάδα μας λοιπόν θα ήθελε μια προσέγγιση που να σέβεται την επικουρικότητα ε, και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στην δημοπράτηση συχνοτήτων Ελπίζουμε επίσης τα κράτη-μέλη να έχουν ισχυρότερη αρμοδιότητα για τη, στον εντοπισμό των ε, αναγκών ε, που θα προκύψουν για τις συχνότητες αυτές. Θεωρώ πως ε, η συζήτηση στο Συμβούλιο δείχνει αυτήν την τάση ήδη και αυτήν την επιθυμία. Τώρα, όπως είπα και χθες όταν συζητούσαμε για την φορητότητα, οι νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εμείς, πρέπει να προσέξουν να μην ε, πέσουν σε ε, λάθη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, να μην εμποδίσουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να, ε, να επιζητούν την ανάπτυξη και να μην υπάρχουν περιορισμοί περιορισμοί και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον περιορισμό ε, σε κατερχόμενη ζεύξη μόνο στις ε, νέες επικοινωνίες. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ο εισηγητής κατέβαλε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί πρόοδο σε αυτήν την έκθεση, κάτι που δεν ήταν σίγουρα εύκολο δεδομένου του τεχνικού χαρακτήρα του ζητήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας για τη δουλειά που έκανε ε, και επίσης προσθέτω ότι στις βασικές του επισημάνσεις συμφωνώ. Θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι το θέμα δεν είναι τεχνικό. Υπάρχει αυτή η τεχνική βάση, αλλά αν ήταν μόνο τεχνικό δεν θα ερχόταν στην Επιτροπή μας. Επομένως έρχεται στην Επιτροπή μας και σε αυτό συμφωνώ Επικουρικά σας λέω ότι είμαι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, είμαι μηχανικός και επομένως μπορώ να το πω όσο αφορά την τεχνική άποψη. Εν πάση περιπτώσει έρχεται στην Επιτροπή μας γιατί. Γιατί να γνωμοθετήσουμε. Ξεκινώ λοιπόν και λέω και εγώ τη γνώμη μου, διότι οι συχνότητες σε όλο τους το φάσμα, αξιοποιήσιμο ή μη αξιοποιήσιμο σήμερα, είναι δημόσια περιουσία, είναι δημόσιο αγαθό, είναι δυνατότητα. Δεν είναι προϊόν, είναι δυνατότητα η συχνότητα. Επομένως, η διαχείρισή του από εθνικές αρχές, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το εξασφαλίζουν αυτό ότι ε, η διαχείριση μέσω των διαφόρων εταιριών που εκπέμπουν άλλοι σε ε, τηλεοπτικά δίκτυα, άλλοι σε ασύρματη τηλεφωνία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετούν ή τουλάχιστον να μην αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον και δεύτερο όσο αφορά τους καταναλωτές των προϊόντων τους, να είναι και ποιοτικά τα αποτελέσματα και φτηνά. Αν αυτή είναι η αρχή, και νομίζω αυτή είναι η αρχή και γι' αυτό το συζητάμε εδώ, πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις έτσι όπως ε, διατυπώνονται από την Επιτροπή, αλλά και η δική μας η δουλειά από την άποψη της γνωμοδότησης. Γι' αυτό είπα ότι σε αρκετά σημεία που υπερασπίζονται έστω και έμεσα αυτό το θέμα, ε, ε, είμαι σύμφωνος δυο τρει ακόμα παρατηρήσει που θέλω να πω. Θέλει να προσέξουμε με αυτή την έννοια σε αυτόν τον ανταγωνισμό που υπάρχει στου παρόχου διαφόρων υπηρεσιών, είτε είναι ψηφιακή τηλεόραση, είτε είναι ραδιοφωνία, είτε είναι ασύρματη ε, τηλεφωνία, όπου παίζουν και ζητούν περισσότερο περιθώριο στις συχνότητες, εμείς, ε, εμείς λέω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό υπέρ του ενός και του άλλου, διότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα κριτήρια νομίζω της δικής μας ε, γνωμοδότησης πρέπει να είναι η υπεράσπιση, όπως είπα, των προηγουμένων, ε, ε, της προηγούμενης κατάστασης. Δεν θα, θα ήθελα, βεβαίως ο εισηγητής μας ίσως, μάλλον προτείνει το αντίθετο, αλλά αν είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί τέτοια βιασύνη για αυστηρές προθεσμίες, δεν το έχω καταλάβει, Φαίνεται πιο λογικό μια προσαρμογή. Ναι, ναι, εντάξει. Το, ναι, το... Ναι, ναι, ναι, το, το κατάλαβα. Και δεύτερη ερώτηση, εντάξει, για να μας βοηθήσει και στον προβληματισμό. Ε, και δεύτερο, επειδή ορισμένε χώρε, όπω αναφέρεται, όπω είναι γνωστό, έχουν ήδη δημοπρατήσει αυτέ τι συχνότητε, τι εμπειρία υπάρχει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, θα μα βοηθούσε η Κομισιόν να κάνουμε και εμεί πιο εύστοχε παρατηρήσει. Με τι παρατηρήσει, ξαναλέω, του εισηγητή μα συμφωνώ, δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω. Θα δω και εγώ τις δικές μου ε, τροπολογίες. Είπα την οπτική με την οποία βλέπω το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Uh, just think for the interpreter... Ναι. Υπάρχει κάποιος ε, θόρυβος. Δεν ξέρω αν είναι κάποια παρεμβολή, διότι ενοχλεί λίγο στα ακουστικά. Ε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, αναφερθήκατε κύριε Χοντή στην Επιτροπή και όντως έχουμε εκπρόσωποι της Επιτροπής ε, να το δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έτυχαν κάποιες ερωτήσεις και θα ήθελα να απαντήσω και να διασκεδάσω και κάποιες από τις ανησυχίες ίσως που εκφράσατε και ο συντάκτης της νομοδότησης αλλά και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι και το διαδίκτυο αλλά και τα οπτικοακουστικά μέσα έχουν μια πολιτιστική διάσταση. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από την έκθεση Λαμή, η οποία δηλώνει ότι δεν είναι οικονομικά προ πολιτισμό, αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα συγκεράσουμε ώστε να βγουν όλοι κερδισμένοι. Υπ' αυτήν την έννοια, πολλά από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση Λαμή, ε, τα έχουμε και εμείς στην πρότασή μας. Παρεπιπτόντος, και η επιλογή της ευελιξίας ήταν ε, τμήμα της έκθεσης Λαμή και να σας εξηγήσω και γιατί ίσως. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Το αν χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, ε, περισσότερο σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες όπως καλωδιακή τηλεόραση ή δορυφορική τηλεόραση. Σε ορισμένες φορές λοιπόν είναι αρκετά χαμηλή, ε, είναι 5% σε άλλες είναι πολύ υψηλό και λαμβάνει το 90% του μεριδίου των συχνοτήτων. Και αυτό φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, όταν ε, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να παρέχουμε κάποια ελαστικότητα στα κράτη-μέλη. Αν δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία, τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φάσμα το οποίο δεν χρειάζεται για τις ε, τηλεοπτικές μεταδόσεις. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ε, ε, συχνότητες αυτές ε, για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, όπως είπε και ο στέκτης της νομοδότησης. Επίσης, αυτοί που δεν το χρειάζονται αυτό το φάσμα συχνοτήτων, πρέπει να έχουν και αυτοί κάποιες δυνατότητες. Είναι κάτι που ανέφερε και ο κύριος Λούερ, η ευελιξία αυτή πρέπει να υπάρχει αν δεν παρέχουμε αυτή την ευελιξία και πούμε ότι είναι μόνο για downlink, χάνουμε μια ευκαιρία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη διεθνή, την διεθνή διαδικασία τυποποίηση. Ε, τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα συμβούν όλα αυτά και αν δεν εκφράσουμε εμεί την άποψή μα για το τι επιθυμούμε, θα συνεχίσουν αυτοί, θα καθοριστούν τα πρότυπα, θα αναπτυχθεί ο εξοπλισμό. και αν εμείς αποφασίσουμε να συνεχίσουμε να μελετάμε το θέμα τη ευελιξίας για κάποια χρόνια, μέχρι να τελειώσουμε μπορεί να υπάρχει ήδη ο εξοπλισμό. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ε, ένας παγκόσμιος κλάδος. Εάν εμείς ε, παρουσιάσουμε κάτι καθυστερημένα, δεν θα ληφθεί υπόψη ε, στη διαδικασία τυποποίησης και κατασκευής του εξοπλισμού και αυτό λοιπόν θα είναι από εκεί και πέρα εις βάρος της Ευρώπης. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ε, θα υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία, θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή του link μας το επιτρέπει και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το άλλο ερώτημα είναι γιατί βιαζόμαστε τόσο να τα επιβάλλουμε όλα αυτά ε, για την προθεσμία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ε, τεχνολογία 4G της κινητής τηλεφωνίας, αλλά αυτό το οποίο ε, εξελίσσεται τώρα, η πέμπτη γενεά, το 5G. Έχουν καθορίσει ήδη τα πρότυπα. Ξέρουμε ότι κάποιες άλλες περιφέρειες έχουν προχωρήσει. Η Κίνα, για παράδειγμα, η κινέζικη κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει η εμπορική χρήση των υπηρεσιών 5G το 2020 και η Ιαπωνία θα χρησιμοποιεί το 2020 υπηρεσίες 5G για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως υπάρχουν πράγματα να εξελίξει. Αν θέλει λοιπόν η Ευρώπη να ηγείται στα θέματα του 5G πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αυτό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το 2020 είναι πολύ σημαντική ημερομηνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να αποτελεί πρόκληση για κάποια κράτη-μέλη. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν δυνατότητες ε, να ε, δοθούν αποζημιώσεις οι οποίες ε, συνάδουν και με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε μια υπόθεση στη Γαλλία ήταν πρόταση για αποζημίωση σε καταναλωτές για αλλαγές που έγιναν. Αυτά μπορούν να γίνουν, συνάδουν με τους κανόνες για κρατικές ενισχύσεις και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας ώστε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε ώστε αυτά τα πράγματα να γίνουν εγκαίρως. Έχουμε τέσσερα χρόνια στη διάθεσή μας μετά την πρότασή μας που σημαίνει αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν όλα αυτά και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκάις, δεκτές παρατηρήσεις σας. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να δώσουμε και μία απάντηση η οποία να μην χάνει και την ισορροπία και να έχουμε και προστασία ενός μοντέλου το οποίο θα προστατεύει και τους καταναλωτές αλλά και το σύστημα κατανομής των ε, ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Ε, θα ακούσουμε και την άποψη του εισηγητή και μετά θα ε, το συζητήσουμε και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Ο κύριος Μαούλου θέλει να απαντήσει. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερως για την αλληλεγγύη ε, που επέδειξαν για την ε, τοποθέτηση της ε, γνωμοδότησης. Όπως είπατε, δεν πρόκειται απλώς για ένα αυστηρά τεχνικό ζήτημα για την χρήση νέων τεχνολογιών και την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια κατάλληλη εξέλιξη. Ε, θεωρώ ότι πρόκειται πρωτίστως για ένα πολιτικό ζήτημα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καθήλυνα αρμόδια για να διασφαλίσει ε, τι γίνεται με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, για πάρα πολλές χώρες. Σας είπα ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτιστικές δυνατότητες, δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στην αρχική μου παρέμβαση. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, κυρίως όσον αφορά αυτή τη διάσταση του 5G και νομίζω όμως ότι η έκθεση Λαμή, την οποία αντικειμενικά θεωρώ ότι αποτελεί σημείο αναφορές για, ε, για τη γνωμοδότησή μου, εγγυάται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η δυνατότητα να έχουμε και αυτή τη διετή παράταση πέραν του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν στρατηγική σημασία τομέα κατά την απόψή μας και να μπορέσουμε να παρέχουμε και στην ε, κινητή την εφορνία το κατάλληλο περιθώριο για να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι μέχρι τις 2 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι πρέπει να καταθέσετε τις τροπολογίες σας Καλή δουλειά στον συνάδελφο Μαούλου και στους κοιόδης ηγητρές. Να ευχαριστήσω και την συνάδελφο από τη Γραμματεία που θα αναλάβει το θέμα. Με αυτό λοιπόν νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι σαν διάφορα. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 30 Μαΐου, 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή για την παρουσία σας. Καλημέρα σας.